Okay, colleagues. we'll start the meeting. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε την συνάντησή μας. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση αυτή που είναι πολύ αργά όπως έχετε παρατηρήσει, άρα όσο νωρίτερα τελειώσουμε, τόσο γρηγορότερα θα φύγουμε. Και εμείς και οι διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε λοιπόν στην έγκριση του θέματος 1 της ημερησίας διάταξης. Ωραία. Περνάμε στο θέμα 2. Όπως γνωρίζετε σήμερα θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση την Επιτροπή Ξέρετε ότι έχουν υποβληθεί 217 τροπολογίες. Ο εισηγητής μας κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες για να επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Πραγματικά εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά, καθώς και η γραμματεία μαζί του και είμαι σίγουρος ότι θα είναι ιδιαίτερα καρποφόρες οι συναντήσεις μας. Παρακαλώ, έχετε εσείς το λόγο, κύριο Δέντα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την υποστήριξή σας συμπεριλαμβανομένου και του εισηγητή. Θα πρέπει να πω ότι ήταν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό θέμα, αλλά πιστεύω ότι η σημερινή ψηφοφορία της έκτασης θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενα και θα μας βοηθήσει στο να καταλήξουμε σε θετικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πριν να περάσουμε <coughs> στην ψηφοφορία Μπορούμε να ελέγξουμε εάν λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψήφι υπέρ. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 24 ψήφισαν, 21 υπέρ, 2 κατά, 2 εποχές, 1 κατά, 2 εποχές. Ωραία, το σύστημα είναι εντάξει. πακέτο συμβιβασμού και, και έχω και μία πρόταση να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Συμφωνείτε όλοι να κάνουμε, να ψηφίσουμε μία φορά για όλες τις τροπολογίες σας. Ναι, τροπολογία συμβιβασμού που έχετε στο φακελό σας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε λοιπόν τον συμβιβασμό 130 όλα... 142 184, 198, 148, 208 και όλες οι άλλες προτάσει προτάσεις τροπολογίας αποσύρονται. Ψηφίζουμε λοιπόν για το πακέτο ε, συμβαστικών προτάσεων. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι σαφές. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 2 κατά, δεν υπάρχουν αποχές. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ήταν εξαιρετική η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Καταλήξαμε σε έναν εξαίρετο συμβιβασμό. Έχουμε μια άλλη ψηφοφορία. Ωραία. Έχουμε και μία άλλη ψηφοφορία. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και κάτι άλλο. Τελική ψηφοφορία στη γνωμοδότηση, στο σύνολό τη, όπω έχει τροποποιηθεί. Έναρξη ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. 23 υπέρ 2 δεν υπήρξαν αποχές και πάλι έχουμε την πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέντε για τη θαυμάσια δουλειά που κάνατε. Θα δώσουμε τώρα την γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ίντε. Κάτι στις, ε, στα διάφορα. Αν όχι, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Μία σύντομη συνεδρίαση μετά τη σκληρή εργασία του εισηγητή και του σκιώδου εισηγητή.